και άλλοι συνάδελφοι βέβαια που δεν ανήκουν στην κοινοπολιτεία. Να εκφράσουμε την ε, τιμή μας για ε, αυτή την εξέλιξη. Την... Σε ευχαριστούμε που ο Ναι, πράγματι. Έχετε δίκιο. Και θα το σημειώσουμε και στα πρακτικά για τη Βασίλη Ελισάβετ. Λοιπόν, να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση. Υπάρχουν κείμενα, έχετε λάβει όλα αυτά τα κείμενα, υπάρχουν αντιρρήσει. Αν δεν υπάρχουν, περνάμε σε μια ανακοίνωση από το Συμβούλιο. Έχω